Δούλικα. Κυρίες και κύριοι, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αμαρφευόρισμων Επενδύσεων πρόκειται να είναι ένα νέο όχημα, τόσο ώστε να μπορέσουμε να ελκύσουμε ιδιωτικές επενδύσει στην οικονομία. Οι μακροπρόθεσμε επενδύσει είναι ένα βασικό εργαλείο, τόσο ώστε να μπορέσει να πάρει το σωστό δρόμο η ευρωπαϊκή οικονομία, μια βιώσιμη ανάπτυξη σύμφωνα με τη στρατηγική για το 2020, το ώστε να μπορέσουμε να έχουμε υψηλή απασχόληση αλλά και υψηλή ανταγωνιστικότητα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενο από τι ε, προσπάθειε που έπιασαν τόπο, ώστε να αποφύγουμε τη γάλυψη των κερδοσκόπων, τόσο ώστε να μπορέσει τώρα να, να καλυφθεί η στρατηγική του 2020 για απασχόληση και κοινωνική πολιτική. Με αυτή την έκθεση θα έχουμε πολύ θετικά αποτελέσματα αποτελέσματα γιατί τώρα θα καλυφθεί η πραγματική οικονομία των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης με αυτή την ε, ε, με αυτή την προσπάθεια θα καλύψουν τους μικροεπενδυτές, θα υπάρχει προστασία τους ακριβώς όπως έχουμε ε, αυτή την διαδικασία της έγκαιρης ε, Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε εμείς πολύ κύριε Φουντσούλη. Μαριάς. Κύριε κύριε πρόεδρε το βασικό πρόβλημα της σύγχρονης οικονομικής λειτουργίας είναι η χρηματιστικοποίηση financialisation της οικονομίας και η λειτουργία μιας οικονομίας καζίνο η οποία επενδύει σε παράγωγα και χρηματιστικά προϊόντα και όχι στην πραγματική οικονομία. και αυτό γίνεται επειδή τα κεφάλαια αποκομίζουν υπερκέρδη για τον λόγο αυτό τρισεκατομμύρια κεφάλαια κυκλοφορούν και αλλάζουν χώρες και χέρια σε λίγες ώρες ενώ οι στρατιές των ανέργων και η παγκόσμια φτώχεια αυξάνεται. προκειμένου να σταματήσει αυτή η κατάσταση απαιτείται σε πρώτη φάση η θεσμοθέτηση μιας νέας glass steagall act η οποία να απαγορεύει στις τράπεζες να είναι βασικός μοχλός της οικονομίας καζίνο μια νομοθετική πράξη που να διαχωρίζει τις εμπορικές από τις επενδυτικές τράπεζες. μόνο έτσι θα μπορέσουν να υπάρξουν κεφάλαια για μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε υποδομές και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. ευχαριστώ. ένα πριν από 2.300 χρόνια ο Μένανδρος είχε δηλώσει ότι τα δάνεια δούλου τους ανθρώπους ποιεί. Και ύστερα από 400 χρόνια ο Πλούταρχος το είπε με πιο σκυρή γλώσσα. Το δανείζεσθε της παραφροσύνης και της μαλακίας εστίν. Η κρίση του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου στην Ελλάδα έπληξε θανάσιμα τη χώρα μας. Ξεζούμισαν το λαό, του άρπαξαν οτιδήποτε για να σώσουν τις τράπεζες. Η ανεργία, ο υποσιτισμός, το κλείσιμο των επιχειρήσεων, τα καταστήματα, η μετανάστευση νέων, οι αυτοκτονίες είναι το σημερινό πρόβλημα της χώρας μας. Αυτά τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια πού θα δοθούν στις τράπεζες ή στο λαό. Γι' αυτό αφήστε τον ελληνικό λαό να κανονίσει τις τύχες του όπως αυτός θέλει. Σας ευχαριστώ κύριε Γκρέζου. Ο κύριος Κέλλη. Äh, Είναι πολύ καλή αυτή η πρόταση που έχει να κάνει με τα ευρωπαϊκά ταμεία μακροπρόθεσμων επενδύσεων. Σιγά σιγά βγαίνουμε από την οικονομική ύφεση. Είναι λοιπόν σημαντικό ως εκ τούτου να δούμε και αυτό το θέμα πλέον, των μακροπρόθεσμων δηλαδή επενδύσεων, ιδίω ε, εκεί που οι επενδύσεις θα είναι αποφελείς προς όλους τους πολίτες. Αυτό το οποίο πρέπει τώρα λοιπόν να μας απασχολήσει είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε αυτές ε, τις βιομηχανίες, σε αυτούς τους κλάδους πρέπει να επενδύσουμε, όπως βέβαια και στον τουρισμό. Πολλά μπορούμε να κάνουμε για να προωθήσουμε την ανάπτυξη μέσω των επενδύσεων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κέλλη. Κύριε Πρόεδρε, ξεκινώ συγχαίροντας τον εισηγητή και τους κύριους εισηγητές που προσπάθησαν να βελτιώσουν τον καρονισμό του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου αλλά δεν μπορώ παρά να διερωτώ με μια και χρησιμοποιήθηκε πολλές φορές ο όρος μικρομεσαίες επιχειρήσεις διερωτώ με μπορούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε αυτή τη χρηματοδότηση Και θα είναι τα ίδια κριτήρια αυτά που θα αξιολογήσουν την ε, δυνατότητα χρηματοδότηση. Γιατί αυτό έχουμε δει στο παρελθόν να συμβαίνει. Πρέπει σε αυτό το Ταμείο των Επενδύσεων να προβλεφθεί ειδικό χώρο, ειδικό κονδύλιο για τι μικρομεσαίες επιχειρήσει. Διαφορετικά, για άλλη μια φορά θα μείνουν εκτό χρηματοδότηση. Μέχρι τώρα το κόσμο όπως και άλλα ταμεία για τις, για τις ε, μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν τέτοια κριτήρια που τις αποκλείουν από τη χρηματοδότηση. Ελπίζω κυρία Επίτροπε να βρείτε μια λύση. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Γκραπίνη. Κανονικά όποιος απουσιάζει την ώρα που και το όνομά του χάνει την ευκαιρία να μιλήσει. Ο κύριος Γουαλτιέρη όμως είχε βγει για λίγη ώρα έξω και έτσι... Μάλλον ο κύριος Βέρ είχε βγει για λίγο έξω και έτσι του δίνω το λόγο για να μιλήσει με τη διαδικασία Καριστιάη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή κύριο Λαμασούρ που έκανε εξαιρετική εργασία. Εγώ υποστηρίζω την θέση του ότι οι επενδύσεις δεν ακολουθούν την βελτιούμε, τους βελτιούμενους οικονομικούς δείκτες στην Ευρώπη. Εάν θέλουμε να στηρίξουμε το σχέδιο Juncker θα πρέπει να προωθήσουμε τις μακροπρόθεσμες ευρωπαϊκές επενδύσεις. Κάτι τέτοιο θα είναι πολύ θετικό γιατί θα οδηγήσει σε περισσότερες επενδύσεις για σημαντικά σχέδια και προγράμματα όπως είναι οι υποδομές που είναι πολύ σημαντικές για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα για χώρες όπως η Σλοβενία που αντιμετωπίζει σοβαρή έλλειψη υποδομών και έχει ε, επίσης προβλήματα για την ανανέωση και, ε, τον, και τη συντήρηση των οδικών δικτύων. Ε, πιστεύουμε πως κάτι τέτοιο λοιπόν θα ενισχύσει την ευρωπαϊκή οικονομία που δεν βασίζεται πλέον μόνο στις τράπεζες. Ευχαριστώ. Ολοκληρώνεται η διαδικασία Καριστιάη. Η Επίτροπος Βεστάιερ έχει το λόγο. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για τα σχόλιά σας. Ε, βέβαια, εμείς από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είμαστε δεσμευμένοι ε, υπέρ της διαθεσιμότητας αυτών των κονδυλίων για μακροχρόνιες επενδύσεις, το συντομότερο δυνατό, γιατί πολλοί είπατε ότι τώρα χρειαζόμαστε τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις συνεργαζόμαστε με τις αρχές ε, των αγορών και των αξιογράφων ώστε να εξασφαλίσουμε κανόνες εφικτούς, εφλιπτούς ε, ώστε να εφαρμοστεί στην πράξη το κείμενο που συζητείτε σήμερα και βέβαια ελπίζουμε και βασιζόμαστε και στην συνεχή συνεργασία μαζί σας για να επιτύχει το όλο εγχείρημα. Ολοκληρώνοντας, να πω ότι το Ταμείο των Μακροπρόθεσμων Επενδύσεων είναι από τα συγκεκριμένα μέτρα που παίρνουν για να έχουμε μια πραγματική ευρωπαϊκή αγορά κεφαλαίου αγορών. Θέλουμε διαφοροποιημένη νέα αγορά δυναμική για να μπορέσουμε να στηρίξουμε την πραγματική οικονομία για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, για να μπορεί να ανθίσει η οικονομία. Γι' αυτό και δημιουργήσαμε ένα στέρεο πλαίσιο που θα παρέχει βεβαιότητα στους επενδυτές ότι δηλαδή θα ε, μπουν τα κεφαλαιά τους στην πραγματική οικονομία σε έργα, σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, σε μεγάλες επιχειρήσεις που θα λάβουν πλέον την τόσο απαραίτητη χρηματοδότηση. Να μπορούν να βασιστούν δηλαδή σε αυτό το κεφάλαιο, μακροπρόθεσμα. Και όπως είπατε πολύ αυτό είναι ένα συμπληρωματικό μέτρο. Έχουμε τη δανειοδότηση από τις τράπεζες, δημόσια κονδύλια και άλλα κονδύλια. Βέβαια θα υπάρχουν και περιορισμοί, διότι ο κανονισμός απαγορεύει επενδύσεις σε τρίτες χώρες που θεωρούνται υψηλού κινδύνου ή μη συνεργατικές δικαιοδοσίες από την χρηματοοικονομική ομάδα δράσης και θα πρέπει ε, και η σύμβαση του ΩΣΑ για το κεφάλαιο και τα εισοδήματα να ε, εφαρμοστεί. Επίσης έχουμε και το Ταμείο και τους κανονισμούς ε, για τις ευρωπαϊκές εταιρείε και εταιρική σχέση. Και αυτό πρέπει να τον λάβουμε υπόψη στον κανονισμό και τις σχετικές διατάξεις. Τέλος, όπως πολύ έχετε κάνει, θέλω και εγώ να ευχαριστήσω τον εισηγητή κύριο Λαμασού και τους σκιώδες εισηγητές που έχουν και αυτή προσιλωθεί στην προσπάθεια να γίνει μια πραγματικότητα αυτό το ταμείο και να μπορούμε να βασιζόμαστε σε αυτό ήδη από τώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Βεστάιερ. Για να ολοκληρωθεί η συζήτηση ο, ο συνάδελφος κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εξαιρετικές ε, καταληκτικές παρατηρήσεις της ε, Επιτρόπου. Θέλω να ευχαριστήσω και όλους τους συναδέλφους που μας υποστήριξαν, ιδίως τους κοιόδες συγητές, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ιταλική Προεδρία που πολύ, πολύ αποφασιστικά και ε, θετικά ολοκλήρωσε τον ε, διάλογο. Αυτή η ποσόστοση το 60% ε, μπορεί να μην πέρασε ως μέτρο, αλλά ίσως να είναι καλύτερο αυτό, διότι δεν έχουμε 60 αλλά 100% πλέον επενδύσεων για ευρωπαϊκά project, για ευρωπαϊκά έργα. Ε, ο συνάδελφος δεν είναι εδώ αλλά ούτε και η κυρία Ματίας στην οποία θέλω να πω ότι με αυτά τα μακροπρόθεσμα κονδύλια δεν θα έχουμε την οικονομία καζίνο, γιατί υποτιφοβάται μια τέτοια οικονομία, το αντίθετο. Θέλουμε τα χρήματα εκεί που υπάρχουν να τα αξιοποιήσουμε και να τα αφιερώσουμε για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση. Ο κύριος Μονό, αν ήταν εδώ και αυτός θα του έλεγα, για να τον καθισχάσω και αυτόν, ότι αντίθετα με αυτά που φοβάται και ανέφερε, οι τράπεζες ιδίως στη δική μας χώρα, τη Γαλλία, συνέχισαν να χρηματοδοτούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τους ρυθμούς των προηγουμένων ετών. Δεν αρκεί όμως αυτό για την ε, εκ νέου όθηση στις επενδύσεις. Ολοκληρώνω με μία σύσταση προς τα κράτη-μέλη. Είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να τα κάνουμε λίγο ελκυστικά, ε, να μην ποσέξει αυτά τα ταμεία. Δηλαδή ε, να είναι η αποταμίευση η πιο φορολογικά ευνοϊκή να δώσουμε δηλαδή κίνητρα για να μπορέσει ε, αυτό το ταμείο να λειτουργήσει. Και νομίζω ότι και η σημερινή συζήτηση έδειξε πόσο χρειαζόμαστε ένα τέτοιο ταμείο. Ευχαριστώ κύριε Λαμασού. Ολοκληρώνεται η συζήτηση.